Honorable members. Πρόεδρος. Βουλευτές θα Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. θα ήθελα λοιπόν να ξαναξεκινήσουμε τις ε, εργασίες μας. Οι δύο σημαντικότεροι βουλευτές ε, του έχουμε την, ε, το σύνδεσμο με την ΕΦΣΑ και την υπεύθυνη των συντονιστών. Σήμερα προβλέπεται η ανταλλαγή ε, απόψεων με τον Δ. Μάρκ Σπρέγγια και ε, δυστυχώς βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ο κύριος Σπρέγγια είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Και πρέπει να πω ότι τον τελευταίο καιρό είχαμε εδώ κοντά μας και άλλους συναδέλφους δικούς σας, οι οποίοι μας είπαν ε, ποια είναι ακριβώς τα φλέγοντα θέματα. Διότι οι οργανισμοί είναι σημαντικοί για μας, καθότι στους ε, οργανισμούς ε, στηρίζετε εσείς τις δικές μας τις πράξεις και ασχολείστε με την εφαρμογή των αποφάσεών μας. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε μια αντίδραση για το τι εκρεμεί ακόμα και περιμένουμε ε, βέβαια την εισήγησή σας ε, για να τεθούν κατόπιν οι ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Σπρέγγια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας δώσω μια γενική έποψη των βασικών μας δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων την περσινή χρονιά. Επίσης, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια και για το μέλλον, για το χρόνο. Αλλά να δούμε και πιο μακρόπνο το μέλλον. Οπότε επιτρέψτε να ξεκινήσω με τις δραστηριότητες ε, του οργανισμού μας, του ECDC. Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες επίση έχουν καθοριστεί για τον χρόνο ε, ε, να αναβαθμίσουν τα εργαστήρια και συνεργασία με τις χώρες διεύρυνσης και επίσης να εξαλείψουν τις ανισότητες τομέα της υγείας. Έτσι θα έχουμε αυτές τις προτεραιότητες και, και για τον χρόνο. Τώρα, όσον αφορά την ε, ε, διεύρυνση, συνεργαστήκαμε ήδη με την Κροατία φέτος και πήγε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε με την Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Όσον αφορά τους μαγουλάδες. Συνεχίζουμε και έχουμε ξεσπάσματα αυτή της ε, ε, ασθένειας στην Άνοιξη Φερρυπίν, στο Λίβερπουλ, στην Αγγλία. Είχαμε τη χειρότερη επιδημία μαγουλάδων από τη δεκαετία του 80. Είχαμε ε, περίπου 200 200, 200 ανθρώπους οι οποίοι αρρώστησαν και, και 40 παιδιά τα οποία μπήκαν στο νοσοκομείο. Και σε όλη την Ευρωπαϊκή συνολικά είχαμε μικρότερο αριθμό συμπτωμάτων και το 2011 αναφέρθηκαν περισσότερο από 30.000 ε, περιπτώσεις. Και μέχρι το 2012 έχουμε ξεπεράσει τις 5.000. Ακόμα πάντως βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά. Και ε, ο στόχος μας είναι ε, μηδενικές, μηδενικές περιπτώσεις, αλλά σε σχέση με τα πρόσθετα χρόνια δεν τα πήραμε τόσο άσχημα. Τώρα, σε σχέση με το 2006 θα δείτε ότι ανεβοκατεβαίνει η επίδοση των μαγουλάδων, αλλά τα πράγματα του ότι είναι ήρεμα φέτος δεν σημαίνει ότι θα είναι το, το ίδιο έτσι ήσυχα και του χρόνου. Οπότε τώρα ερχόμαστε να δούμε στο γιατί και οι ανισότητε στην υγεία αλλά και οι μαγουλάδες είναι προτεραιότητες πολιετής για μας. Εάν πρόκειται να εξαλείψουν τους μαγουλάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο 95% κάλυψη από ε, εμβόλια σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις κοινότητες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό η κάθε χώρα ξεχωριστά. Οι δε ευρωπαϊκέ χώρε, τι χώρε τη Ένωση με υψηλή κάλυψη, ακόμα ε, ε, πλήσονται από το φαινόμενο γιατί έχουμε ε, κάποια γειτονική χώρα που μεταδίδει την ασθένεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να εξαλείψουμε το φαινόμενο χωρί να μιλήσουμε για τι ανισότητε. Ακόμα και εκεί που έχουμε μεγάλη κάλυψη, τότε έχουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε μη ε, καλυπτόμενη πληθυσμία Και αυτή είναι η μετανάστες, είναι η Ρωμά και άλλοι μη προνομιούχοι. Και εκεί πέρα η, η κάλυψη από τα εμβόλια είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σαν, ε, ε, σαν, αποτέλεσμα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτές τις χώρες. Και γι' αυτό στο Δουβλίνο την περασμένη μήνα συναντηθήκαμε με ειδικού από τα κράτη-μέλη, με εκπροσώπους των Ρωμά και με εκπροσώπους των τράβελων, των περιπλανωμένων. Σε, αυτό το, σε αυτή τη συνάντηση συμφωνήθηκαν 10 ε, προτάσεις για το πώς οι χώρες είναι δυνατόν να αυξήσουν την κάλυψη από τα ε, εμβόλια σε, στις ευάλωτες ομάδες και στον γενικά τροπληθισμό. Τώρα θα, αυτές τις προτάσεις θα τις παρουσιάσουμε στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, συνάντηση της σχετική για την ανοσοποίηση των ε, ανηλίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω όσον αφορά τα ε, εργαστήρια τι έχει γίνει. Οπότε είχαμε επίσης ε, φαινόμενα ε, ηλαράς, πρώτη για ηλαρά διαφθούν και όχι για μαγουλάδες τον περασμένο μήνα. Και αυτό ήταν μια καινούργια εμπειρία και για όλες τις υπηρεσίες και την ΕΦΣΑ και τη δική μας υπηρεσία. Για αυτό το, τον, ε, τον, την, διαδικασία ταχείας αποτίμησης του κινδύνου. Είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον όμως ότι πήγαμε σε συντονισμό όσον αφορά την χρήση ε, των δοκιμών των εργαστηριακών για σαλμονέλα. Οπότε είχαμε ε, ασθενείς σε διαφορετικά κρατημέλη οι οποίοι είχαν μολυνθεί από σαλμονέλα ε, συνήθως έφταιγε γι' αυτό ε, κρέας γαλοπούλας. Ε, πρόκειτο για πάρα πολύ επιτυχή επομένως συνεργασία για τα εργαστήρια και αυτό θα μας ε, θωρακίσει για το μέλλον. Βεβαίως, φέτος θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιδρούμε καλύτερα όσον αφορά ε, ασυνήθιστα, προσδόκητα συμβάντα. Είχαμε ας πούμε πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά για ένα νέο ιό που λέγεται κορώνα και μοιάζει πολύ με του, την οικογένεια ιών, την κατηγορία ιών που ονομάζουμε SARS. Οπότε, έχει αυτό να κάνει και με το AIDS και με την έμπολα. Είναι συγγενείς. Οπότε θα έπρεπε κάτι να κάνουμε μέσα σε το Σαββατοκύριακο. Και παράλληλα είχαμε στις κάτω χώρες, ε, στη Ηνωμένο Βασίλου και στη Γερμανία, ε, τα εργαστήρια τα οποία και από τη Γενική Διεύθυνση Κομισιόν και από την υπηρεσία μας είχαν ε, χρηματοδοτηθεί, οπότε προχώρησαν εργαστηριακά σε δοκιμές για αυτό το νέο ιό. Και έγινε επομένω αποτελεσματική συνεργασία χωρίς επικάλυψη των προσπαθειών. Στις 9 το βράδυ την Κυριακή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με την υπηρεσία μας σε σχέση με, την έγκαιρη προειδοποίηση του σχετικού σύστημα της ε, ανταπόκρισης σε αυτά τα γεγονότα και υπήρχαν πληροφορίες για αυτές τις νέες εργαστηρικές δοκιμές. Την ιδέα τη Δευτέρα ξεκινήσαν οι, σε όλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να να μελετούν το πώς θα υπάρχει βέβαια περισσότερες πληροφορίες παντού και κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο σωστός τρόπος ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε τους, δεδομένου, δεδομένους, τους περιορισμένους πόρους σχετικά τη δημοσία υγεία όταν έχουμε επομένω μια κοινή ε, απειλή τότε θα πρέπει να εργούμε με τέτοιο τρόπο και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια αφετηρία σίγουρη ε, και έτσι είναι δυνατόν να συντονίζεται και να αντιδρά σε απειλές που ανακύπτουν ε, μέσω της Επιτροπής ε, Ασφάλειας της Υγείας. Τώρα, σας παρακαλώ, θα ήθελα λίγα λεπτά για να σας μιλήσω για τα σχέδια που έχουμε το 2013 και πέρα. Έχουμε πάρα πολύ βασικά ορόσημα το 2013, τα οποία πρέπει να σας επισημάνω. Πρώτα-πρώτα, το 2013 θα είναι η χρονιά κατά την οποία θα υλοποιήσουμε και θα εφαρμόσουμε μια νέα ενισχυμένη πολιτική όσον αφορά την επιστημονική ανεξαρτησία. Έτσι θα επικυροποιήσουμε και θα ε, επεκτείνουμε το έργο που ήδη ε, επιτελούμε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να άρουμε και να προλάβουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων. Δεύτερον, πρόκειται να έχουμε συνεχή αξιολόγηση εξωτερικών ε, ανεξαρτήτων αξιολογητών. Θα έχουμε αξιολογητέ επίση από φέτο για την συλλογή των δεδομένων και θα έχουμε επομένω την ε, τελική έκθεση του 2013 και θα εγκρίνουμε το στρατηγικό προγραμμα πρόγραμμα 2014-2020. Ξεκίνησε η προπαρασκευαστική εργασία. Τον περασμένο μήνα δε στη Στοκόλμη είχαμε αυτή τη, την κοινή συνάντηση στρατηγική όπου ήρθαν ε, ε, υψηλού επίπεδου εμπειρογνώμες από τα κράτη-μέλη ε, και συμμετέσχε και το, το συμβουλευτικό μας φόρουμ και έτσι μπορέσαμε να έχουμε πραγματικές συνεισφορές και έτσι καταλήξαμε σε ένα έγγραφο διαβούλευσης με τους ε, συνομιλητές μας. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό από αυτές τις συζητήσεις με τους ε, συναδέλφους στα κράτη-μέλη ήταν ότι θέλανε συνέχεια και συνέχιση επί της ουσίας όσον αφορά το έργο της υπηρεσίας μας. Όμως, ε, ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε θα μεταβληθεί και αυτό βεβαίως σχετίζεται με το ότι θα υπάρχουν λιγότεροι πόροι και είναι αλήθεια ότι στον τομέα της υγείας θα πιέζει το ελληνικό προπολογισμό. Νομίζω όμως ότι μπορεί να πετύχει περισσότερα με λιγότερο πόσο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας, ευχαριστώ και την κυρία Γιούτα Χάου, την εισηγήτρια για τον προπολογισμό ε, για τη βοήθειά τους. Να σας δώσω όμως άλλα δύο ε, παραδείγματα αλλαγής. Πρώτα-πρώτα, τι κάνουμε όσον αφορά τα δεδομένα της ε, έρευνας ε, όσον αφορά τις ε, μολυσματικές ασθένειες. Τα πράγματα θα αλλάξουν μέχρι το 2020 και θα πρέπει να έχουμε σε πιο, με πιο φιλικό τρόπο στην ε, συλλογή των δεδομένων και υπάρχει και κάποια εφαρμογή στα smartphone μέχρι τότε. Όμως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα, στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα, τη μικροβιο, τα μικροβιολικά εργαστήρια και έτσι θα τους βοηθήσουμε να γίνει συντονισμός και να έχουν και στα κράτη-μέλη νέες τεχνολογίες για τη δημοσία υγεία και αυτό να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο ε, ε, αν το 2020 να είμαστε καλά, ακόμα μπορώ να έρθω εδώ στην Επιτροπή σας και τότε θα μιλούμε για την ε, αντιμικροβιακή αντίσταση, για το AIDS, για την ε, φυματίωση, τη γρήπη, τις ε, προετοιμασία για πανδημίες κλπ. κλπ. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να νομίζω θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε όλες τις απροσδόκητες απειλές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω πώς και πώς τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπρέγκερ για την εισήγησή σας. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιανακουδάκη που είναι η, ε, η σύνδεσμός μας με την υπηρεσία σας. Σας ευχαριστώ κύριε Σπρέγγερ γιατί ήταν πολύ ενημερωτικά τα όσα μας εξηγήσατε. Βεβαίως και ε, είναι απογοητευτικό ότι δεν έχουμε περισσότερους συναδέλφους να σας ακούσουν αλλά πάντως ε, είναι γνωστό ότι έχουν μια επιθετική στάση προς τις περιφερειακές ε, ε, ε, υπηρεσίες. Θεωρώ ότι περισσότερο δεν έχουν λόγο ύπαρξης, όμως επί του προκειμένου νομίζω ότι κάτι θα βγει, θα είναι χρήσιμο, θα βοηθήσει όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο σας. Οπότε γι' αυτό και το τίμιο σύνδεσμος με χαροποιεί και είναι η μόνη υπηρεσία δική σας την οποία επιθυμούσα ανέκαθεν να, να κάνω αυτή τη δουλειά Ήρθε σε επαφή με τον Μάρκ και με την ομάδα του, οπότε είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο ε, για να μπορέσουμε να εκπροσωπηθούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο πέρασε κάποιος καιρός και τώρα αυτό το οποίο θέλουμε είναι το ότι θα έχουμε τακτές συναντήσεις με τους εκπροσώπους πριν πάνε στις ε, συνεδριάσεις ε, οπότε να μπορούμε να περάσουμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου σε αυτούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει προσθέμενη αξία από όλες τις υπηρεσίες. Πάντως εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερος το ότι η υπηρεσία σας ήδη έχει κάνει μεγάλες εξορμίες δαπανών σε δύο τομείς. Από ό,τι βλέπω εδώ, πρώτα-πρώτα ε, τον προϋπολογισμό του 2013 όσον αφορά την εποπτεία, 13% 30% πόσο έχετε κόψει. Τόσο πολύ καλό είναι αυτό το που κάνετε και επίσης ε, όσον αφορά αποστολές και συναντήσεις και εκεί είχε κάνει οικονομίες. 60.000 ευρώ εξοικονομήσατε. Συγχαρητήρια προς τον Μάρκ και προς ε, το επιτελείο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Τώρα ένα άλλο τομέα πάρα πολύ σημαντικός όπου η υπηρεσία σας ε, αποδίδει είναι το τι έγινε με αφορμή τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Ευρωπαϊκού 2012 που ήταν ε, αιτίε, πλατφόρμες τέλο πάντων να μεταδοθούν κάποιες ασθένειε. Μια που μετακίνητο ο κόσμος για να δει τα γεγονότα αυτά, να τα παρακολουθήσει. Οπότε μεγάλη μα χαρά η υπηρεσία σας. είχε κάποιε ε, πάγιες ε, εκθέσεις συνεχώς κάθε μέρα για τις ε, ασθένειες τι γίνονταν στην Ευρώπη και αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται στα κρατη οπότε όλοι προσέχανε για το τι αρρώστιες κυκλοφορούν. Τώρα ένα πρόβλημα που πρόκειψε πέρυσι εκτός από το πρόβλημα του Διευθυντικού Συμβουλίου ήταν η αναδιοργάνωση, η στελέχωση του προσωπικού και από εκεί πρόκειψε το εξή. Όποτε κάνει κανεί αναδόμηση και μετακινεί τον κόσμο γύρω-γύρω, ε, άλλοι θα είναι ευχαριστημένοι και άλλοι θα παραπονιούνται. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι ε, λίγοι θεώρησαν ότι έχουν αδικηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι προέκυψε για τίποτα το πολύ βαρύ. Και τελικά η αναδιοργάνωση οδήγησε σε αποδοτικότερη λειτουργία. Δυστυχώ το Κοινοβούλιο α, ακόμα δεν έχει ασχοληθεί με το πρόγραμμα όσο θα έπρεπε, ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο δυναμικοί και να δούμε μήπως κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να μου πούν πώς βλέπουν τα πράγματα και ένα δε από τα προβλήματα που συνάντησα και τα συζήτησα με τον πρόεδρό μας είναι η σχέση μεταξύ εμού ως συνδέσμου και άλλων συνδέσμων που ασχολούνται με άλλες υπηρεσίες. Γιατί υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους θα πρέπει να συνεργαστούμε, να έχουμε τόσο κοινά κριτήρια και να μπορούμε να ωφελθούμε όσο είναι περισσότερο αυτές οι υπηρεσίες. Άρα, περισσότερο συντονισμός. Ίσως, ε, έτσι, να, να, οι σύνδεσμοι να συναντιόμαστε κάθε 6 μήνες. Να συζητούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι καλύτερε πρακτικές, όμως αυτό είναι θέμα του Προέδρου. Του χρόνου θα γίνει μια επίσκεψη στην Στοκχόλμη, περιμένω πώς και πώς, να πάω εκεί, να μιλήσω στο προσωπικό, σε όλα τα τμήματα της υπηρεσίας και θα σκόπιμο να πάνε άλλοι φέτος σε σχέση με πέρσι, τόσο ώστε όλοι να μάθουν τι γίνεται. Αυτά. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λίντα Μακάου. Όπω είπε και η κυρία ε, Γιανακουδάκη, κρίμα που δεν είναι εδώ άλλοι συνάδελφοι. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ συντονιστών. Είμαι ευγνώμη για τι πληροφορίε που δόθηκαν για την Ιλαρά. Πέρσι το συζητήσαμε το θέμα. Ποιε είναι οι τάσει, έχουμε μόνο αριθμού. Είπατε για το Split και για το Liverpool. Η τάση ποια είναι. Αυξητική, ελέγχεται η κατάσταση, μειώνονται τα κρούσματα. Τι συμβαίνει. Ε, τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, λαμβάνονται τα μέτρα, τα κατάλληλα να καταλαβαίνουν πως σημαντικός είναι ο εμβολιασμός οι γονείς. Επίσης, υπάρχουν οι ευάλωτες κοινωνίες, όπως είπατε, ή τα άταμα τα οποία όντως δεν κατανοούν πολύ καλά τα μηνύματα περί δημοσίας υγείας. Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, στο Guardian, διάβαζα για τις ασθένειες τις οποίες μεταδίδουν αυτοί που ταξιδεύουν σε εξωτικά μέρη και φέρνουν κάποιους ιούς από την Αφρική ή αλλού που εμφανίζονται για πρώτη φορά. Τροπικές ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν. Υπήρχαν στην Ολλανδία και στις ΙΠΑ ε, κάποια κρούσματα τέτοιων ασθενειών ε, από την Αφρική. Διερωτώ με, στοχεύουμε και προς αυτά τα άτομα οι μετανάστες από τις χώρες αυτές οι οποίοι ξαναγυρίζουν στις χώρες τους, περνούν διακοπές και ξαναφέρνουν άλλους. Ε, είναι ευάλωτοι κατά κάποιο τρόπο, ίσως όχι απαραίτητο οικονομικά διότι ταξιδεύουν σε τέτοιες χώρες εξωτικές, αλλά εν πάση περιπτώσει φέρουν στην Ήπειρό μας ασθένειες τις οποίες, ε, οι οποίες μας βρίσκουν απροετοίμαστος, δεν είμαστε έμπειροι γι' αυτά. Και τελευταία ερώτηση, η οικονομική κρίση μιλήσαμε για την υγεία, για τις ε, ε ανισότητες. Μάθαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Υπάρχει περίπτωση άλλων πανδημικών ασθενειών. Πώς βλέπετε εσείς να επηρεάζει η οικονομική κρίση την δημόσια υγεία, τα προγράμματα εμβολιασμού και άλλα τέτοιου θέματα. Ευχαριστώ. Κύριε Σπράγγελ, μήπως μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την κυρία Γιανακουδάκη για τα ευγενικά της σχόλια. Ε, Χρήστος, σας στο Λονδίνο, ανταλλάξαμε πώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς κυρία Μακιούν για τις ερωτήσεις σας. Η Λαρά είναι μία ασθένεια σαν τυφώνας. Πηγαίνει ανά την Ευρώπη, ταξιδεύει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κρούσματα στη Ρουμανία ένα χρόνο. Την επόμενη χρονιά ήταν η Γαλλία και είδαμε πρόσφατα ότι επίσης υπήρχε πρόβλημα με την Ιλαρά στην Βόρεια Αγγλία. Βεβαίως όλα εξαρτώνται από τον εμβολιασμό ή μη ατόμων τα οποία είναι ιδιαίτερα ε, ευάλωτα. Και υπάρχουν διακυμάνσεις στην Ιλαρά. Κάθε τέσσερα χρόνια βλέπουμε να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα κρουσμάτων. Τώρα, φέτος βλέπουμε να έχουν μειωθεί τα κρούσματα σε σχέση με πέρσι. Όχι διότι όλοι κάναμε καλά δουλειά μας, όχι διότι είναι Μεγαλύτερο αριθμό των εμβελιαζόμενων, αλλά είναι θέμα εξάπλωσης του ιού. Είναι πολύ σημαντικό να εμβολιάζονται οι άνθρωποι. Δεν είμαι όμως πολύ αισιόδοξο, διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι αντίθετοι στον εμβολιασμό που θα ήθελαν να δημιουργήσουν ε, φήμες για το τις απειλές των εμβολίων. Υπάρχουν και κοινότητε και έχουμε στη Γερμανία διάφορα παραδείγματα με την Ρούντολφ Steiner Σούλε, τη σχολή αυτή, όπου λέγεται ότι υπάρχει συγκέντρωση μη εμβολιασμένων ατόμων. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί έχουμε αύξηση τη ηλαράς. Τώρα, η Ρωμά, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Ε, εκλήθην από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία. Είχα με τους κάποιους Ρωμά συναντήσεις. Είναι μια πάρα πολύ ε, είναι μια κοινωνία που διαφέρει από τη μία περιοχή στην άλλη. Είδα κάποιους mediators όπω λένε, κάποιους μεσάζοντες, πώς να τους πω, οι οποίοι βοηθούν κάπω την κατάσταση και είδα με ευχαρίστηση ότι πολλοί από αυτούς που θέλουν να προωθήσουν τα θέματα υγείας κάποια στιγμή σπουδάζουν και γίνονται γιατροί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κάθε κοινότητα να παρέχει τέτοιε υπηρεσίε δημόσια υγεία. Αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι ότι η κοινότητα των Ρώμα δεν είναι κατά του εμβολιασμού. Απλώ δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση και δεν είναι οι λύσεις που τους προτείνονται πάντα στα μέτρα τους. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας για τις εξωτικές ε, και τροπικές ασθένειες, αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Πρόσφατα, στη Μεγάλη Βρετανία είδαμε ότι ένας ασθενής είχε αιμορραγικό πυρετό και εντυπωσιάστηκα από τις δημόσιες υγειονομικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο που μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν και υπάρχουν σύνδεσμοι και δεσμοί με το εξωτερικό και προσπαθούν να ιχνηλατήσουν τις ε, νόσους αυτές τις ε, παράξενες και τους ασθενείς διότι αν κάποιος επίσης ασθενήσει ε, σε μια εξωτική χώρα ας πούμε και γυρίσει στην πατρίδα του δεν θα μεταδώσει αυτό το νιό ή το νόσημα σε άλλους. Τώρα, κάποιος ασθενής σε ένα αεροπλάνο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να πρέπει εμείς να αξιολογήσουμε αν μπορεί να έχει κολλήσει, να έχει μεταδώσει το πρόβλημα, την ασθένειά του στους άλλους συνταξιδιώτες. Τώρα η Λετζιονέλα είναι, ε, είναι πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια, αλλά έχουμε καλά συστήματα για να ανοιχνεύσουμε τα προβλήματα που ενδεχομένως ε, μπορούν να πλήξουν ξενοδοχεία. Τώρα, όσον αφορά την ε, οικονομική κρίση. Εμένα με επασχολεί το θέμα αυτό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Βεβαίως, διότι ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα πέσουν στην ανεργία και ίσως θα δούμε αύξηση περιθωροποιημένων και ευάλωτων ατόμων στην κοινωνία. Ε, αλκοολικών ή άλλων. Και όλοι αυτοί μπορούν να είναι και πιο ευάλωτοι στην φυματίωση και στο AIDS. Συγχρόνως όμως βλέπουμε αύξηση αυτών των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία και συγχρόνως καλύτερα μέσα για βασικές ε, φροντίδες υγιεινής. Αυτό το οποίο είδαμε τελευταία στην Ελλάδα είναι να υπάρχει εξάπλωση του ε, ιού μεταξύ των πολιτών που ήταν οροθετική. Εάν δεν έχει κανείς χρήματα για θεραπεία υποκατάστασης. Εάν δεν έχει χρήματα για ανταλλαγή υγειονομικών προγραμμάτων, υπάρχει καταστροφή. Η καταστροφή δεν θα έρθει ούτε αύριο, ούτε τον επόμενο μήνα, αλλά ίσως του χρόνου. Αυτό συμβαίνει, αυτή, αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι πρέπει για τα προγράμματα αυτά να αφιερώσουν κάποια κονδύλια. Ξέρουμε επίσης ότι αυξάνεται η αντιμικροβιακή αντίσταση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν επίσης Υπάρχει επίσης το θέμα της μεταφοράς ασθενών από μια χώρα για ένα νοσοκομείο σε άλλη. Εάν και είναι πολύ σημαντικό το screening. Εάν δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, βλέπει να υπάρχει αντίσταση ε, στα μικρόβια. Τώρα, για τη φυματίωση. Αυτό ε, μας ε, απασχολεί και η αντίσταση σε μεγάλο αριθμό φαρμάκων ε, στον ιό της φυματίωσης μας απασχολεί και ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη στελέχη τα οποία δεν μπορούμε ακόμη να θεραπεύσουμε. Άρα δεν ξέρουμε ε, ποια είναι η σωστή θεραπεία έγκαιρα για το κάθε ασθενή. Δεν ξέρω εάν συνειδητοποιείτε ότι η θεραπεία της φυματίωσης φτάνει στα ποσοστά μόνο 50% και πολλοί τελικά πεθαίνουν από φυματίωση. Άρα υπάρχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την οικονομική αυτή κρίση. Πολύ ωραία κύριε Σπρέγκερ. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τα θέματα αυτά στην Επιτροπή μας, δηλαδή τι είδου επιρροή άσκησε η χρηματοπιστωτική κρίση στη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, όσον αφορά στα δημόσια συστήματα υγείας, ε, στη χρηματοδότησή τους, ε, στην ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Όταν υπάρχει μια περίπτωση κατά πόσον κάποιος θα πάει σε ένα νοσοκομείο και στην περίπτωση αυτή πρέπει να περάσει μέσα από τομογράφο, θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη χρηματοδότηση. Γιατί αν δεν είναι γνωστό μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε, αλλά τελικά αυτό που παίζει ρόλο είναι ε, να ε, επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτών των προβλημάτων. Βλέπω ότι ήρθαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κανείς το λόγο. Αν όχι, ε, θα ήθελα εγώ να κάνω μια στάνταρτ ερώτηση. Η στάνταρτ ερώτηση που γίνεται είναι τι κάνει ο δικός σας οργανισμός όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Διότι <clears throat> το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Παρόλα αυτά θέλουμε σε έναν τέτοιο οργανισμό να έχουμε τους καλύτερους. Ε, και αυτό το αίτημα είναι πάντα και δικό μας. Επιθυμούμε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Ε, πολλοί εμπειρογνώμονες όμως ε, δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους και γι' αυτό ερωτώ ο δικός σας οργανισμός τι κάνει ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει και νομίζω ότι ενδιαφέρει και όλες τις ομάδες. Παρακαλώ. Χαίρομαι πολύ που ελκύει την προσοχή σας το θέμα μας. Βεβαίως και είμαστε σε επαφή με ένα σωρό εμπειρογνώμονες και ειδικού. Βέβαια. Ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις ε, οικονομικών συμφερόντων από το δικό μας προσωπικό. Από εκεί ξεκινήσουμε λέμε γιατί αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια κοινή προσέγγιση και από την εμπειρία μπορώ να σας πω ότι είναι κάπως κινούμενος στόχος. Πριν από δύο ώρες μόλις, το ελληνικό συνέδριο έδωσε μια συνέντευξη τύπου για αυτά, για την σύγκρουση συμφερόντων. Θα διαμορφωθεί μια συνένεση για το πώς θα προσεγγίσουν το θέμα, αλλά ακόμα και έτσι, ακόμα και έτσι, ακόμα και από τώρα προσέχουμε πάρα πολύ το τι γίνεται προκλούμε από κοντά, το προσωπικό που ασχολείται με την γρήπη, ε, τους περνά από χίλια κόσκινα αυτούς που μπαίνουν στα πάνελ και ένας συμπρογνώμονας μπορεί να μην αντιμετωπίζει σύγκρουση φορών αλλά εάν πάει να δουλέψει για μια φαρμακευτική εταιρεία, τότε θα τον βγάλουμε από την Επιτροπή Συνοπεργαζόταν. Σας λέω, προσέχουμε το θέμα πάρα πολύ. Και ελπίζουμε ότι τον επόμενο μήνα θα εγκριθεί η στρατηγική μας, αλλά επίσης θα κάνουμε και μια γενικότερη προσέγγιση, οπότε θα λάβουμε υπόψη και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. και όποτε επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας θα σας τα δείξω όλα αυτά από κοντά οπότε θα διαπιστώσετε από κοντά πώς χειριζόμαστε το θέμα. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία θα δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για τα θέματα τα οποία τέθηκαν κατά τη συζήτηση και ιδιαίτερω θα αρχίσω με το θέμα του εμβολιασμού, το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα. Απλώ να αναφέρω ότι η Επιτροπή σε συνεργασία με την Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε κάποια συμπεράσματα να αφορά τον παιδικό εμβολιασμό. Και εκ των υστέρων θα οργανώσει την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν μία διάσκεψη για να δει ποιε είναι ενδεχομένω οι πρωτοβουλίε που θα μπορούσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λυθούν ώστε να ενθαρρυνθούν όλε οι χώρε να καλύψουν πλήρω τι ανάγκε παιδικού εμβολιασμού. Βεβαίω, για, τις, ε, για το ξέσπασμα πολλών κρουσμάτων ερυθράς ε, που είναι επίγον πράγμα επίσης πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεύτερη παρατήρηση αφορά σύσταση του Συμβουλίου που βασίζεται στο άρθρο της συνθήκης περί δημοσίας υγείας, όπου πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο ε, για να υπάρξει γενικότερος εμβολιασμός. Και υπάρχει έκθεση ε, που αφορά τα άποψη των διαφόρων κρατών μελών, θα δημοσιευτεί από το Συμβούλιο και θα δείτε κατά πόσον έχει εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη αυτή η σύσταση που έπρεπε να εφαρμόσουν. Αυτή τη στιγμή, από όσων ξέρουμε, είναι μεικτά τα αποτελέσματα. Τρίτο στοιχείο που αναφέρεται αφορά την πανδημίες και την πανδημικό εμβολιασμό μετά από την πανδημία του 2009 της γρήπης, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προετοιμάσει ένα μέσο, ένα μηχανισμό για δημόσιες αγορές εμβολίων. Δηλαδή, αντί να αγοράζει κάθε χώρα εμβόλια χωριστά και να διαπραγματεύεται με τις φαρμακοβιομηχανίες, είπαμε ότι από κοινού κάποιες χώρες θα διαπραγματεύονται μια κοινή σύμβαση για την αγορά αυτών των εμβολίων. Και ίσως όπως είδατε, χθες Είχαμε την έκθεση του κυρίου Παρνιού, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή σας και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία συμπεριλάμβανε και η ε, νομική, ε, νομικού περιεχομένου πρόταση Επιτροπής. Προχωρούμε λοιπόν ε, προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να έχουμε μια κοινή σύμβαση μεταξύ ομάδων κρατών που θα αγοράσουν από κοινού τα εμβόλια για όλους. Αυτό επίσης έχει σχέση με την πρωτοβουλία διασυνοριακής ε, λήψης μέτρων και εδώ στην περίπτωση του πανδημικού, του γενικού εμβολιασμού και θα αφορά διάφορα ιατρικά προϊόντα. Όπως ξέρετε η Επιτροπή σα ενέκρινε την έκθεση αυτή, θα πάει στην Ολομέλεια, συζητείτε σε προηγμένο επίπεδο και το όλο θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο θα ενισχύσει την σχέση μεταξύ του ε, αξιολόγηση κινδύνου και αντιμετώπιση του κινδύνου από το κέντρο. Βεβαίω, δεν θα πρέπει μεταδοτικέ ασθένειε με άλλου τύπου ασθένειε να συγχέονται, αλλά προ το μου προχωρούμε καλά. Ο κύριος Σπράγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του κέντρου μας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παραγωγική στον τομέα αυτό. Χθες παρακολούθησα επί μία διάσκεψη για τον εμβολιασμό κατά της γρήπης, όπου είχαμε εκπροσώπους της βιομηχανίας Πληρώσαμε εμείς όμως το ειστήριό μας για να παρακολουθήσουμε τις εργασίες τους. Και θέλω να αποσφυρίσω το εξή. Αφενός, καλό είναι που υπάρχει η σύσταση του Συμβουλίου για τον εμβολιασμό ομάδων κινδύνου. Απ' την άλλη είναι πολύ σημαντικό η φαρμακοβιομηχανία να επομιστεί τις ευθύνε τη, ώστε να προσφέρει το καλύτερο δυνατό εμβόλιο. Και είναι σαφές από κάποιες μελέτες που έγινε από το κέντρο μας ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Είναι λοιπόν σημαντικό να αποσαφινιστεί ότι και εκείνοι έχουν ένα μέρος ευθύνης να επομιστούν. Δεν ξέρω αν μπορώ εγώ να εκφράσω την απόψή ε, μου για την πρωτοβουλία ε, της διασυνοριακής ε, ε, συνεργασίας όταν υπάρχει κίνδυνος αλλά βλέποντας τις συζητήσεις που κάνατε χθες, νομίζω ότι είναι θετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ε, πράγματι, εχθές ε, πετύχαμε μια πολύ καλή συμβιβαστική πρόταση και ε, όσον αφορά την έκθεση που αναφέρατε, καλή είναι η συμβαστική πρόταση που επιτεύχθηκε στις συζητήσεις, στις δημόσιες συζητήσεις γίνονται πολλές αναφορές ε, στον οργανισμό σας. Ε, αφού το είπε και η Σκιώδη Εδώ μπορούμε να προβάλλουμε την υπεραξία, γιατί τελικά μόνο μία υγεία έχουμε όλοι μας και τα 500 εκατομμύρια. Και αν μπορεί κανείς να προστατεύσει καλύτερα αυτήν την υγεία, εργαζόμενος πέρα από τα σύνορα, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και εδώ ε, μπορούμε να προβάλλουμε την ευρωπαϊκή υπεραξία. Εμείς ε, το δουλεύουμε αυτό καθημερινά. Εσείς βέβαια ελέγχετε την εργασία αυτή. Εσείς είσαστε αρμόδιος στη Στοκχόλμη, στον οργανισμό σας ε, και εσείς ε, μας λέτε κατά πόσον σε ορισμένα θέματα ε, θα πρέπει να επανέλθουμε ή όχι. Λέτε βέβαια ότι είσαστε ανεξάρτητοι. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μερικές φορές καλύτερη επικοινωνία με τους ανεξάρτητους αυτούς οργανισμούς. Δεν βλέπω κανείς να ζήτησε περαιτέρω το λόγο. Κατόπιν τούτου ευχαριστώ εκείνους ε, οι οποίοι ήρθαν σήμερα στην Επιτροπή μας και εκείνους που δεν ήρθαν, αυτούς που δεν ήρθαν θα τους ενημερώσουμε στο μέλλον, στις συνεδρίες των συντονιστών, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται στο μέλλον ε, τέτοιου είδους ε, συζητήσεις. Και δεν πρέπει να επιπλήττουμε αυτούς που ήταν εδώ. Αυτοί που δεν ήταν εδώ έχασαν. Κύριε Σπρέγκερ, σας εύχομαι τα καλύτερα και τον Απρίλιο του επόμενου έτους θα σας επισκεφτούμε στη Στοκχόλμη και θα μπορέσουμε επιτόπου να δούμε τι ακριβώς κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας. So, und wir sind damit auch schon am Ende der... Τελειώσαμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Γιατί εχθές ακυρώσαμε τα υπόλοιπα, τα σημεία 20 και 21, τα εξετάσαμε εχθές. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συναντηθούμε στις 5 και 6 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι έκατσαν εδώ μέχρι το τέλος και ε, σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό ταξίδι στις πατρίδες σας για όσους θα επιστρέψουν.